Liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζω θερμά. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχουμε τις ε, δηλώσεις του Συμβουλίου για την παρουσίαση του προγράμματος ε, της Τσεχικής Προεδρίας. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω θερμά.